οι προσκεκλημένοι μας μπορεί να προσεγγίσουν πολύ διαφορετικά το θέμα. Γι' αυτό λοιπόν διοργανώσαμε αυτή τη συνεδρίαση πάνω στο θέμα πυρηνική ασφάλεια στην Τουρκία και στην περιφέρεια της χώρας αυτής. Εδώ θα στηριχθούμε και στα ε, μέσα προσχώρησης και γι' αυτό ε, μετέχει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία σε μεγάλο βαθμό είναι ε, γνώστη των θεμάτων αυτών και μετά την προσχώρηση της Βουλγαρίας πριν από λίγα χρόνια. Και αναφέρομαι σε τέσσερις αντιδραστήρες οι οποίοι σε αυτή τη φάση μπορεί να παρουσιάζουν κάποιους κινδύνους και οι μέθοδοι οι οποίοι προβλέπονται για την προστασία του πληθυσμού σε περίπτωση ατυχήματος ίσως να μην έχουν ξεκαθαριστεί. Η Τουρκία σκοπεύει στην κατασκευή τριών εγκαταστάσεων. Η μία είναι στο Ακουγιού, η πιο γνωστή. Έχει προβλεφθεί να κατασκευαστεί σε συνεργασία με τη Ρουσία. Η λειτουργική εξέταση του προγράμματος είναι υπό εξέταση. Η ρωσική πλευρά έχει ήδη διαπραγματευτεί με μια τουρκική επιχείρηση και υπάρχει επίσης πέραν του Ακουγιού και ένα σχέδιο για τη Μαύρη Θάλασσα στη Συνόπη στο βόρειο τμήμα δηλαδή της Τουρκίας και αυτό θα γίνει μαζί με την Νότιο Κορέα σε συνεργασία. Βέβαια το θέμα αυτό μπορούμε να το δούμε μέσα από διαφορετικά πρίσματα, να δούμε γενικά το θέμα της πυρηνικής ενέργειας ως οικολόγος πράσινος θα έλεγα να το δούμε μέσα από αυτό το πρίσμα το ζήτημα που μας απασχολεί. Μπορούμε να το δούμε και μέσα από τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του θέματος και το ζήτημα της ευθύνης της Τουρκίας απέναντι σε γειτονικέ χώρες. Υπάρχουν ε, διεθνείς συμβάσεις που θα πρέπει να μελετηθούν μετά από το Τσερνομπίλ και τη Φουκουσίμα. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα για τους γείτονε, γιατί τέτοιου είδους ζητήματα συνεπάγονται αναλήψη ευθυνών και προς ανθρώπους που μένουν στην ευρύτερη περιοχή. Επίσης είναι το θέμα των ενεργειακών επιλογών και πηγών. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία δεν χρησιμοποιεί πυρηνική ενέργεια, αλλά περιβάλλεται από άλλες χώρες που το κάνουν όπως η Αρμενία, που είναι πολύ κοντά γεωγραφικά. Ε, ε, είναι ε, κοντά στην Τουρκία. Έτσι λοιπόν δεν έχει καθόλου πυρηνική ενέργεια η Τουρκία τώρα. Οι πόροι στις εναλλακτικές πηγές δεν γίνονται αντικείμενο εκτετάλευση σε καμία περίπτωση λοιπόν. Η συζήτηση έχει ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό θα συνδεθούμε με Skype για, με μια κυρία η οποία είναι μέλος της Greenpeace, Greenpeace και εκπρόσωπος των οργανώσεων των τοπικών εναντίον της οικοδόμησης ε, του ακουγιού. Τώρα πώς θα γίνει η σύνδεση τεχνικά, ε, οι εμπειρίες μας με τις τεχνολογίες αυτές δεν είναι πάντα ε, καλές, αλλά εδώ μου λένε ότι τα πράγματα μάλλον θα πάνε καλά. Η επιλογή αυτών των πυρηνικών εγκαταστάσεων ανησυχεί πολλούς. Ξέρετε ότι η Τουρκία παρουσιάζει υψηλούς σεισμολογικούς κινδύνους. Ζητήσαμε λοιπόν από έναν καθηγητή ειδικό των προβλημάτων αυτών να προσπαθήσει να μας διαφωτίσει για τους σεισμολογικούς κινδύνους των περιοχών οι οποίες μας ενδιαφέρουν. Ε, θα έχουμε και τον πρέσβη της τουρκικής δημοκρατίας, τον καλωσορίζω, τον κύριο Κιούνεραλπ. Θέλω να ευχαριστήσω και τον Αντιπρόεδρο κύριο Κουμουτσάκο, ο οποίος είχε την ιδέα αυτής της συζήτησης, πήρε την πρωτοβουλία για την οργάνωσή της και θα του δώσω το λόγο για να μας εξηγήσει για ποιους λόγους θεώρησε να οργανώσει αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και τον ευχαριστώ που το έκανε με απόλυτα ανοιχτό τρόπο. Ευχαριστώ <clears throat> πολύ κυρία Πρόεδρε. Ε, καλημερίζω όλους όσοι συμμετέχουν στη σημερινή συζήτηση. Ο σκοπός ε, της πρωτοβουλίας αυτής ήταν ε, να γίνει μια ψύχρεμη συζήτηση για ένα θέμα <clears throat> ιδιαίτερα ευαίσθητο για ένα θέμα που προκαλεί το ενδιαφέρον, την ανησυχία και τον προβληματισμό ε, πολλών ε, πολιτών, όχι μόνο στη χώρα μου, που είναι μια γειτονική χώρα της Τουρκίας. Το ζήτημα ξεπερνάει ε, τις γειτονικές χώρες. Είναι ένα ζήτημα ευρύτερου ενδιαφέροντος, ένα ζήτημα περιφερειακό και ευρωπαϊκό ταυτόχρονα. Η ευαισθητοποίηση για το ζήτημα που συζητάμε σήμερα βεβαίως πυροδοτήθηκε από τις τραγικές, δραματικές εξελίξεις και γεγονότα, τα πρόσφατα δραματικά γεγονότα στην Ιαπωνία. Πιστεύω λοιπόν ότι η σημερινή ψύχρεμη συζήτηση θα συμβάλλει στο ώστε να δοθούν οι σωστές διαστάσεις στο ζήτημα το οποίο έχει ανακύψει. Θα μου επιτρέψετε να μοιραστώ μαζί σας πολύ σύντομα ορισμένες σκέψεις για το ευρύτερο αυτό θέμα, αλλά και για το ειδικότερο της ε, πυρηνικής ασφάλειας στην Τουρκία. Η πυρηνική ασφάλεια, κυρίε και κύριοι, είναι ένα θέμα που ξεπερνάει αναφυσβήτητα τα σύνορα ενός κράτους. Επομένως, είναι κατανοητό ότι τα σχέδια για την κατασκευή πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγικής σε μια ιδιαίτερα σεισμογενή χώρα, στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι λογικό να παρακολουθούνται με προσοχή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και τους άλλους ευρωπαϊκούς θεσμούς, σύμφωνα άλλωστε με την επίσημη θέση που έχουν πάρει κατά καιρού και αρμόδιοι επίτροποι. Είναι γεγονός ότι η περιοχή γύρω από την πόλη του Ακούγιου βρίσκεται στο νοτιοδυτικό άκρο του ρήγματος της Ανατολίας. Πολλοί σεισμολόγοι έχουν χαρακτηρίσει την ευρύτερη περιοχή ως περιοχή υψηλής σεισμικότητας εξαιτίας των ισχυρών σεισμών που έχει δώσει κατά καιρού το συγκεκριμένο αυτό ρήγμα. Ακόμα όμως και αν δεχτούμε τους ισχυρισμού επιστημόνων, κάποιων επιστημόνων, για μέτρια ή χαμηλή σεισμικότητα της περιοχής, θα ήταν νομίζω λάθος να παραβλέψουμε την γενικότερη σεισμική δραστηριότητα και τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει σε έναν ενδεχόμενο πυρηνικό σταθμό. Εξάλλου σε διεθνές επίπεδο υπάρχουν χαρακτηριστικά παραδείγματα όπου η φύση διέπευσε με τρόπο πανηγυρικό επιστημονικούς χαρακτηρισμούς και επιστημονικά συμπεράσματα. Θα δώσω μόνο ένα παράδειγμα. Στο κόμπε της Ιαπωνίας, που είχε χαρακτηριστεί ως χαμηλή σεισμικότητα. ο ισχυρός σεισμός μεγέθους 7 Ρίκτερ του 1995 άφησε πίσω του χιλιάδες νεκρούς και καταρρεύσεις όλων των κρίσιμων εγκαταστάσεων όπως γέφυρες, κτίρια κλπ. Γενικότερα, σε χώρες με γενικότερη υψηλή σεισμικότητα δεν μπορεί να διασφαλιστεί η μέγιστη ασφάλεια κρίσιμων κατασκευών, ακόμα και αν αυτές βρίσκονται σε περιοχές χαμηλής ή μέτριας σεισμικότητας. Ο πρόσφατος σεισμός και το τσουνάμι στην Ιαπωνία και η πυρηνική τραγωδία που ακολούθησε απέδειξαν ότι όσο σύγχρονες και αν είναι εγκαταστάσεις, όσο αυστηροί και αν είναι κανονισμοί κατασκευής πυρηνικών εργοστασίων, η φύση μπορεί να του ξεπεράσει. Επίσης δεν μπορούμε να παραβλέψουμε και την αντίδραση της κοινή γνώμης, της Τουρκίας αλλά και πολλών κρατών μελών για την κατασκευή ενός τέτοιου ε, εργοστασίου στη συγκεκριμένη αυτή περιοχή. Οι κάτοικοι του Ακούγιου και των γενετικών περιοχών και των γειτονικών περιοχών εκφράζουν συχνά την έντονη ανησυχία τους για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει το πυρηνικό σχέδιο επίσης και στον τουρισμό της περιοχής. Σύμφωνα άλλωστε με μελέτες, η αύξηση της θερμοκρασίας θάλασσας που θα προκαλούσε η δραστηριότητα ενός πυρηνικού εργοστασίου θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμα και σε καταστροφή της θαλάσσιας ζωής στην περιοχή για περισσότερο από 10 χρόνια, ενώ τα κέντρα ψήξης του αντιδραστήρα θα επηρεάσουν το κλίμα στη Μεσόγειο. Σε κάθε περίπτωση, και κλείνω με αυτό, οι μελέτες για την καταλληλότητα της περιοχής του Ακουγιού είναι ένα εξελίξη. Ο Γενικός Διευθυντής της Ρόζατομ, κ. Σάπροφιν, δεσμεύτηκε σε μια συνέντευξη τύπου που έδωσε πρόσφατα στην Άγκυρα, την Τρίτη, ότι θα δεν θα αποκρύψει τίποτα από τους πολίτες και ότι σε περίπτωση αμφιβολιών για την ασφάλεια της περιοχής θα ανασταλούν τα σχέδια κατασκευής του σταθμού. Με αυτές τις σκέψεις και με αυτά τα από πλευράς μου ε, γεγονότα τα οποία παρέθεσα, αλλά και ορισμένες εκτιμήσεις, προσδοκώ και περιμένω μια ενδιαφέρουσα επικοδομητική συζήτηση, βεβαίως περιμένοντας με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τη γνώμη των ειδικών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Euh, Ευχαριστώ τον κύριο Κουμουτσάκο. Θα δώσω το λόγο τώρα στους προσκεκλημένους. Θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Γκιουλκάν. Είστε καθηγητής πολιτικός μηχανικός στο Πανεπιστήμιο της Άγκυρας και είστε πρόεδρος μιας διεθνούς ένωσης για την αντιμετώπιση των συνεπειών των σεισμών Έχετε γνώσεις λοιπόν για τις σεισμολογικούς κινδύνους στις περιοχές της Συνόπης και του Ακουγιού. Έχετε το λόγο. Πρόεδρε, καλή σας μέρα. Χαίρομαι που σήμερα μπορώ να πάρω μέρος στη σημερινή σας συνάντηση και να σας ενημερώσω για τους σεισμολογικούς κινδύνους που παρουσιάζονται στις δύο αυτές περιοχές. Εδώ και 35 χρόνια ασχολούμαι με τις υποθέσεις αυτές. Το θέμα της ασφάλειας από τους σεισμούς είναι κάτι το οποίο θεωρώ πως είναι απόλυτα θεμητό. Όχι μόνο για τη συγκεκριμένη χώρα, τη χώρα μου, αλλά και για τις γειτονικές χώρες και ε, αυτό φάνηκε από τα σχόλια της Προέδρου και τα σχόλια που ακολούθησαν. Πρώτον, θα ήθελα να σας μεταφέρω τους λόγους για τους οποίους η Τουρκία προωθεί την κατασκευή αυτών των μονάδων τα τελευταία 35 χρόνια. Αυτή είναι μια προσπάθεια η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει οδηγήσει σε αυτά αποτελέσματα, όπως κάθε άλλη χώρα που έχει πυρηνικές εγκαταστάσεις και η Τουρκία χρειάζεται να διευρύνει την ηλεκτροπαραγωγή της βάση και να διαφοροποιήσει τις πηγές ενέργειας σε συνδυασμό και με τις υπόλοιπες διαθέσιμες πηγές. Η Τουρκία εξαρτάται από εισαγωγές για την παραγωγή ενέργειας που καλύπτουν τις ανάγκες της βιομηχανικέ. της. Το 65% της ενέργειας που χρειάζεται εισάγεται ουσιαστικά. Οι πρώτες Οι πρώτες τοποθεσίες που έχουν επιλογή, επιλεγεί μου είναι γνωστές. Έχει υπάρξει και μια τρίτη ε, επιλογή προτινόμενη κοντά στη Βουλγαρία, αλλά ως προς αυτήν δεν είμαι απόλυτα ενημερωμένος. Οι δύο λοιπόν πιθανές τοποθεσίες είναι η Συνόπη στο βορρά και το Ακουγιού στο νότο. Η Συνόπη βρίσκεται στην Μαύρη Θάλασσα. Η προσπάθεια για το ακουγιού έχει ήδη ξεκινήσει. Έχουν υπάρξει επίσημες ανακοινώσεις. Οι μελέτες συνεχίζονται όμως. Και θυμίζω ότι για το ακουγιού τα τελευταία δέκα χρόνια δεν έχει υπάρξει κάτι συγκεκριμένο εκτός από μια ενημερωμένη και επικαιροποιημένη μελέτη για τις σεισμολογικούς κινδύνους, τις οποίες την οποία παρουσίασε εδώ και δύο χρόνια. Οι μελέτες για τη Σινόπη έγιναν ανάμεσα στο 2005 και στο 2010, σε μια πενταετή περίοδο. Οι μελέτες του Ακουγιού λοιπόν υπάρχουν, έχει υπάρξει μια άλλη μελέτη εκτός από τη δική μου, για τη θαλάσσια υδροδυναμική της περιοχής. Έχουν υπάρξει 110 μελέτες επιμέρους που καλύπτουν επιμέρους λεπτομερέστερα θέματα. Η σεισμικότητα και ο κίνδυνος που συνδέεται με το επίπεδο αυτό της σεισμικότητας έχει γίνει αντικείμενο μελέτης για αρκετές δεκαετίες. Έχω προσωπικά εμπλακεί στην διεξαγωγή αυτών των μελετών. Κατά τη διάρκεια των μελετών αυτών ακούστηκαν πολλές απόψεις, ακούστηκαν πολλές αντιλήψεις και πολλές εκτιμήσεις για το κίνδυνο. Οι αντιλήψεις αυτές έχουν οριμάσει και πολλές έχουν αλλάξει κιόλας. Σχετικά με την γνωστή δεδομένη σεισμικότητα του ακουγιού, το θέμα έχει ως εξής. Αυτοί οι μικροί κύκλοι δείχνουν το επίκεντρο όπου έχουν υπάρξει σεισμικές δονήσεις. Είδαμε την κατανομή των δονήσεων αυτών. Είδαμε τις γεωγραφικές του συγκεντρώσεις είδαμε τον τρόπο με τον οποίο δημιουργήθηκαν. Και έχουν γίνει και αρκετές μελέτες και σε σχέση με τα βάθια. Εμείς αυτό το οποίο κάνουμε σαν πολιτική μηχανική είναι να προβλέψουμε τι θα γίνει σε μια συγκεκριμένη περιοχή κάποια στιγμή στο μέλλον εάν υπάρξει μια σεισμική δόνηση ενός δεδομένου επίπεδου. θέλουμε λοιπόν εμείς ε, ε, οι συνέπειες αυτές, ε, ακριβώς με όποια μέτρα μπορούμε να πάρουμε, να καταστήσουν τις πιθανότητες επιβεβαίωσης αυτών των ζημιών που θα προβλέψουμε όσο πιο μακρινή, όσο πιο απίθανη σε εισαγωγικά γίνεται. Ε, ξέρετε ότι έχουμε ένα ρήγμα στη συγκεκριμένη περιοχή και βέβαια και οι μελέτες ε, όταν ασχολούνται με την τεκτονική των ε, ρήγματων δεν είναι κάτι το πάρα πολύ εύκολο. Έχουμε τα ρήγματα στο Λος Άντζελες σαν παράδειγμα, είναι ένα από τα πιο γνωστά θέματα και οι μελέτες δεν επιβεβαίωσαν, δεν προέβλεψαν τους τελευταίους σεισμούς στην περιοχή. Όταν εξετάσει κανείς τους ορίζοντες θα ελέγξει, θα δει ότι υπάρχει ε, τον τελευταίο καιρό έλλειψη σεισμικότητα στην περιοχή. Κοιτάξτε, θέλω να προσπαθήσω, δυσκολεύομαι λίγο γιατί θέλω να προσπαθήσω να παρουσιάσω τη συγκεκριμένη μελέτη όσο πιο ε, εύκολη στην κατανόησή της. Δεν θα ήθελα να χρησιμοποιώ λέξεις που ίσως κάθε φορά θα θέλουν εξηγήσει. Βλέπετε εδώ τη συχνότητα ε, των ε, ε, σεισμών ε, σύμφωνα με τη συχνότητα που διαπιστώσαμε μέχρι τώρα όπως την προβλέπουμε τις επόμενες δεκαετίες. Εμείς αυτό το οποίο κάνουμε είναι να προσπαθήσουμε να δούμε τι θα συμβεί στο μέλλον επί τη βάση των γνώσεων του παρελθόντος και επί τη βάση των στοιχείων για τα γεωλογικά χαρακτηριστικά μιας συγκεκριμένης τοποθεσίας στην ουσία αυτό το οποίο κάνουμε είναι παίρνουμε το τι γνωρίζουμε από τα τελευταία 100 χρόνια και κάνουμε μία προβολή των στοιχείων αυτών ας πούμε τα επόμενα 5.000 χρόνια. Βέβαια υπάρχουν πάρα πολλά λάθη και στα στοιχεία που έχουμε και όσο περίπλοκα να είναι και τα στοιχεία τα οποία έχουμε. πάντα έχουμε να κάνουμε με μεγάλα ποσοστά αβεβαιότητας. Ε, έχει υπάρξει αναφορά και για ένα πιθανό ρήγμα πολύ κοντά στο ακουγιού. Αυτό είναι μια πρόταση που έχει γίνει από σεισμολόγους, αλλά έχει αμφισβητηθεί από άλλους εξίσου αξιόπιστους γεωλόγους. Η συζήτηση η οποία έγινε δημοσιεύθηκε και οι απαντήσεις ε, έγιναν σε ένα συγκεκριμένο περιοδικό από έναν Βρετανό γεωλόγο και η γλώσσα η οποία χρησιμοποιείται είναι αρνητική θα έλεγα για την συγκεκριμένη επιλογή. Και πρέπει να αποσυρθεί γενικά η πρόταση. Γιατί τη ε, οι μελέτες ξεκίνησαν αρκετά αργά και ολοκληρώθηκαν πριν δύο-τρία χρόνια. Όλες οι καταμετρήσεις έγιναν γύρω από τις συγκεκριμένες περιοχές για την αξιολόγηση των κινδύνων των περιοχών αρχών. Υπάρχουν και κάποιες άλλες μελέτες για την ευρύτερη περιοχή, στις οποίες όμως εγώ δεν ενεπλάκην προσωπικά το ιστορικό των ε, δονήσεων στην περιοχή ε, ε, περιορίζεται, εγγράφεται θα έλεγα σε ένα πολύ μεγάλο ρήγμα, το βόρειο αν, ε, ρήγμα της Ανατολίας. Είναι κάτι το οποίο σε μέγεθος αντιστοιχεί και στο ρήγμα του Αγίου Ανδρέα στην Καλιφόρνια. Βρίσκεται στο νότο της τοποθεσίας της Συνόπης, και έχουμε ελέγξει μια μεγάλη χρονική περίοδο ε, εμφάνισης τέτοιων φαινομένων. Όπως και στο Ακουγιού έγιναν ε, τρεις μελέτες για την τοποθεσία της συνόπης, για την παρακολούθηση ε, και την καταλογοποίηση των μικροσυσμικών δραστηριοτήτων. Είναι κάτι το οποίο μας δείχνει μερικές φορές το τι θα ακολουθήσει σε επίπεδο σεισμολογικό και βλέπουμε ότι αυτές οι μικροσυσμικές δραστηριότητες εντοπίζονται και περιορίζονται γεωγραφικά στο εσωτερικό της περιοχής η οποία καλύπτεται ε, από το ρήγμα αυτό της Βόρειας Ανατολίας. Εδώ βλέπετε τους σταθμούς ελέγχου τους οποίους αναπτύξαμε στην περιοχή την περίοδο 2007 με 2009. Αναπτύξαμε 12 σεισμολογικούς σταθμούς για 18 μήνες. Και εδώ έχετε το ιστορικό των σεισμικών δραστηριοτήτων έτσι όπως κατανέμεται στην περιοχή αυτή που όπως είπα βρίσκεται πολύ κοντά στο ρήγμα της Βόρειας Ανατολίας και εδώ είναι οι εκτιμήσεις τις οποίες έκανα με τους συναδέλφους, εκτιμήσεις οι οποίες δίνουν μια πρώτη εικόνα της περιοχής. Οι περιοχές που είναι οι πιο σκιασμένες προς το κόκκινο είναι αυτές που παρουσιάζουν υψηλότερες δραστηριότητες και τα υπόλοιπα χρώματα έχουν χαμηλότερα επίπεδα επικινδυνότητας. Αυτές οι εκτιμήσεις μας. Οι εκτιμήσεις μας για τη συνόπη βρίσκονται περίπου στο ίδιο επίπεδο επικινδυνότητας με το ακουγιού. Το ακουγιού και η συνόπη είναι οι πλέον σταθερές περιοχές στην ευρύτερη περιοχή. Σεισμολογικά λοιπόν είναι οι πιο, οι πιο σταθερές περιοχές στο σύνολο της χώρας. Το 1989 υπήρξε ένας μείζον σεισμός στον Άγιο Φραγκίσκο. Στο Λόμα Πριέτο, 110 χιλιόμετρα νότια από την πόλη του Αγίου Φραγκίσκου. αλλά μία από τις βάσεις της γέφυρας που συνδέει την πόλη του Σαν Φρανσίσκο με το Όκλαντ κατέρευσε κατά τη διάρκεια του σεισμού αυτού. Η αντικατάσταση συνεχίζει να βρίσκεται υποκατασκευή. Καταλαβαίνετε ότι αρχιτεκτονικά είναι προκλητική αυτή η γέφυρα, η οποία πρέπει να είναι και αισθητικά ευχάριστη και η οποία βασίζεται σε έναν πυλώνα, ο οποίος θα φέρει το σύνολο του βάρους ε, της ε, γέφυρας η οποία θα είναι επικρεμάμενη και θα φτάνει το μήκος των 130 μέτρων. Η περιοχή βρίσκεται 8 μίλια δυτικά του ρήγματος του Σαν Αντρέα και επίσης στην ίδια απόσταση από ένα άλλο ρήγμα το οποίο ε, είχε δώσει δραστηριότητες σεισμικές το 1937. Υπάρχει λοιπόν ένας πολύ μεγάλο, μια πολύ μεγάλη στήλη, μια πολύ μεγάλη ε, ε, η οποία προβλέπεται να έχει ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα αντοχής σε σεισμικές απειλές, απειλές επίπεδου που δεν προβλέπονται στην Τουρκία. Λοιπόν, επί τη βάση όλων των γνωστών στοιχείων και το ακουγιού και η συνόπη φαίνεται ότι είναι κατάλληλες για την κατασκευή πυρηνικών εγκαταστάσεων. Κατάλληλες. Με αυτό θέλω να κλείσω. Σας ευχαριστώ κύριε καθηγητά Γιούλκαν. Αυτή είναι η γνώμη σας. Θεωρείτε λοιπόν ότι τα δύο σημεία αυτά τα οποία επελέγησαν είναι σημεία μικρότερου σεισμολογικού κινδύνου, μικρότερη σεισμικής έκθεσης. Παρ' όλα αυτά οι καταστροφές τις οποίες γνωρίσαμε τελευταία στον πυρηνικό τομέα δείχνουν ότι υπάρχει μια σειρά συμβάντων που δεν συνδέονται αποκλειστικά με σεισμικές δραστηριότητες. Ξέρετε τι έχει συμβεί στη Φουκουσίμα και τι εξακολουθεί να συμβαίνει. Υπήρξε συνδυασμός συμβάντων που κατέστησε τις πιθανότητες τις οποίες εσείς αναφέρατε πολύ πιο επιβαρυντικές κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες. Και δεν νομίζω ότι το συμπέρασμα σας είναι τέτοιο το οποίο μπορεί να μας καθησυχάσει και σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις που έγιναν στους τοπικούς πληθυσμούς της Τουρκίας φαίνεται ότι η μεγάλη τους πλειοψηφία είναι εχθρική προς την κατασκευή αυτών των εγκαταστάσεων. Θα μιλήσουμε με, τον κύριο, με την κυρία Άτιτσι, η οποία είναι υπεύθυνη για τις περιφερειακές εκστρατείες της Greenpeace. Θα την ακούσουμε από τηλεδιάσκεψη. Ε, η διερμηνία ε, θα δούμε αν θα ακολουθήσει, γιατί στις καμπίνες δυστυχώς δεν ακούμε καλά τους ήχους. Προς το παρόν δεν ακούμε τίποτα στη διερμηνία, στις καμπίνες. Κοιτάξτε, η πρόεδρος λέει, σας διακόπτω γιατί θα πρέπει να προσπαθήσετε να μιλάτε ίσως σε απόσταση σταθερή από το μικρόφωνο, γιατί έχουμε μια φωνή η οποία έρχεται σε μας με πάρα πολλές διακυμάνσεις. Θα μιλήσει αγγλικά λέει η κυρία, αλλά δυστυχώς στις καμπίνες δεν ακούγεται. because um, we have witnessed many uh, uh, misinformations until now from these uh, bodies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 Middle East Technical University. uh They are making researches and uh their findings are that the uh amount of cesium hear me? Vous êtes parti, mais Can you hear me? Oui, oui, oui, on vous entend, on vous entend. Allez. Α, κάποια στιγμή σας χάσαμε, αλλά τώρα σας ακούμε, λέει η Πρόεδρος. Συνεχίστε, κυρία μου. Σας ακούμε. Je n'entends pas. Can you hear me now? Yes. Ça va? Φαίνεται όμως ότι η κυρία δεν μας ακούει. Est-ce que vous nous entendez? Μας ακούτε, ρωτάει η πρόεδρος ε, την κυρία Χιλάλ Ατίτσι.

περιμένουμε από τους τεχνικούς μας να μας πούν εάν μπορούμε να επανασυνδεθούμε με την κυρία, αλλιώς θα προχωρήσουμε στον επόμενο μιλήτη. Θα επανέλθουμε. Αργότερα δεν υπάρχει τεχνικά η δυνατότητα να παρακολουθήσουμε. Θα δώσουμε τώρα το λόγο στον πρέσβη τον κύριο Γιούνερ Αλπ Ευχαριστώ Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Σας ευχαριστώ και σας και τον κύριο Κουμουτσάκο για την πρωτοβουλία της διοργάνωσης αυτής επί ενός πολύ επικέρου θέματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το γνωρίζουμε, αλλά και στην Τουρκία, αφού η πυρηνική ενέργεια είναι αντικείμενο έντονης συζήτησης, η οποία έγινε ακόμη πιο έντονη μετά το ατύχημα στην Φουκουσίμα. Είμαι πολύ ευτυχής ε, από την πρωτοβουλία αυτή και ελπίζω ότι αφού η τουρκική πλευρά της αντιπροσωπείας παρουσιάσει τις θέσεις της, ε, θα συνεχίσουν ε, και μετά ε, οι συζητήσεις και με την ε, νέα, μετά τις εκλογές με τους νέους συναδέλφους. Είναι... Σταματήστε, δεν μπορούμε να ακούσουμε. Υπάρχει μεγάλο τεχνικό πρόβλημα. είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό και επίκαιρο και σε σχέση με το άνοιγμα του κεφαλαίου για την ενέργεια. Εγώ δεν είμαι ειδικό στα θέματα αυτά. Ήδη ακούσαμε την άποψη του ειδικού. Και μετά τη δική μου παρέμβαση θα έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε και την παρουσίαση της Greenpeace. Ε, καταρχήν λοιπόν εγώ θα προσπαθήσω να σας παρουσιάσω τη γενικότερη εικόνα ε, των ενεργειακών θεμάτων. Μετά θα πω δύο λόγια και για την πυρηνική. Το πρώτο θέμα που πρέπει να αναφέρουμε είναι ότι η Τουρκία εξαρτάται απόλυτα από τις εισαγωγές των υδρογονανθράκων το 91% συγκεκριμένα του πετρελαίου και το 98% του φυσικού αερίου που καταναλώνει εισάγονται από το εξωτερικό και συνολικά οι εισαγωγές είναι το 70% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας. Έχουμε υδροηλεκτρική ενέργεια σε μεγάλο βαθμό. Η αιωλική και η ηλιακή ενέργεια, όπως ξέρετε, ακόμα είναι πολύ δαπανηρές και ενώ έχουμε αρκετό δυναμικό για την ανάπτυξη της υδροηλεκτρικής ενέργειας, υπάρχουν βέβαια κάποια περιβαλλοντικά θέματα που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και που μετριάζουν την πλήρη αξιοποίηση των πόρων αυτών. Γνωρίζετε το θέμα αυτό. Αν σκεφτείτε ότι η ανάγκη σε ηλεκτρική ενέργεια προβλέπεται να αυξηθεί κατά 6 με 7% κάθε χρόνο, να αυξάνεται, μετά από την ταχύτατη ανάπτυξη της τουρκικής οικονομίας και αν δείτε επίσης και την αλλαγή του κλίματος σε σχέση με τη χρήση πηγών υδρογονανθράκων σε αυτήν την κατάσταση η πυρηνική ενέργεια για την Τουρκία αλλά και για πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες και άλλες ε, σε όλο τον κόσμο. Η πυρηνική ενέργεια λοιπόν γίνεται μια εναλλακτική που πρέπει να εξεταστεί με πολύ προσοχή και σοβαρότητα. Η οικονομία μας αναπτύσσεται ταχύτατα όπως σας είπα, αυξάνεται επίσης ο πληθυσμός της χώρας και ο συνδυασμός της εξάρτησης από εισαγόμενα ορεκτά καύσιμα και η ανάγκη μείωσης των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα και αύξησης της ενεργειακής ασφάλειας, αυτός ο συνδυασμός κάνει την, διερεύνη, την ε, μελέτη και το, της πυρηνικής ενέργειας ε, μια σημαντική εναλλακτική για πολλούς. Όπως ε, ανέφερε και ο καθηγητής Γκουλκάν, δεν είναι καινούρια αυτή η κατάσταση. Η Τουρκία εξέταζε το ενδεχόμενο ανάπτυξης ε, πυρηνικής ενέργειας εδώ και 35 χρόνια τουλάχιστον. Και από την αρχή ήδη η περιοχή του Ακουγιού ε, είχε προτιμηθεί για τους λόγους που ακούσαμε. Και με τη σύναψη μιας συμφωνίας, κυβερνητικής συμφωνίας με τη Ρωσική Ομοσπονδία, η κατασκευή και λειτουργία ενός πυρηνικού εργοστασίου σε αυτήν την ακτή της Μεσογείου όπου βρίσκεται το Ακουγιού αποφασίστηκε. Είναι το πρώτο έργο σε αυτόν τον τομέα γιατί για πρώτη φορά μια ξένη χώρα θα αναλάβει να, να κατασκευάσει, ε, να ε, είναι ιδιοκτήτη και να λειτουργεί ένα τέτοιο εργοστάσιο σε άλλη χώρα. Βέβαια θα διέπεται κανονιστικά από τις τουρκικές αρχές ε, και νομοθεσία και κανονισμούς και θα υπόκειται στον έλεγχο της ε, Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας στη Βιέννη. Θα χρηματοδοτηθεί το έργο αποκλειστικά από τη Ρωσική Ομοσπονδία η τουρκική εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας αναλαμβάνει ε, να αγοράζει μισή, τη μισή παραγωγή για 15 χρόνια, τη μισή παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από το εργοστάσιο και προβλέπεται επίσης στα πλαίσια της ε, συμφωνίας αγοράς ότι η εταιρεία θα μεταβιβάσει το 20% του κέρδους της στο τουρκικό Υπουργείο Οικονομικών, στο τουρκικό δημόσιο. Θα κατασκευαστούν τέσσερις μονάδες του τύπου VVER 1200, που είναι ένα νέος τύπος μοντέλου και το εργοστάσιο αναμένεται να παράγει Ε, περίπου 4.800 ΜΒ ηλεκτρικής ε, ενέργειας και θα ολοκληρωθεί γύρω στο 2020. Θα υπάρξει μεταφορά τεχνολογίας, ε, περιλαμβάνεται και αυτή η διάσταση στη συμφωνία για το έργο. Οι τουρκικές εταιρείες και Τούρκοι πολίτες θα απασχοληθούν και θα εκπαιδευτούν, καταρτιστούν κατά τη διάρκεια της κατασκευής και λειτουργίας του εργοστασίου. Ε, επίσης έγινε μια διαπραγμάτευση με την Ιαπωνία για την κατασκευή του δεύτερου πυρηνικού εργοστασίου στη Σινόπη, στην περιοχή που ανέφερε επίσης ο καθηγητής Γκουλκάν, αλλά για λόγους που είναι γνωστοί σε όλους μας, οι διαπραγματεύσεις ε, σταμάτησαν, ε, διεκόπησαν μετά το ατύχημα στη Φουκουσίμα και το τσουνάμι. Το ατύχημα αυτό βέβαια έφερε στο φως την ανάγκη για πιο στεναρά και αυστηρά μέτρα ασφαλείας που θα πρέπει να εφαρμοστούν σε όλα τα ε, υπάρχοντα και μελλοντικά εργοστάσια και κατέδειξε επίσης την ανάγκη για βελτίωση της διεθνούς συνεργασίας σε θέματα πυρηνικής ενέργειας. Η Τουρκία, αυτό είναι σαφέστατο, αυτονόητο, θα φροντίσει στον ανώτατο βαθμό να εφαρμόζει κάθε κριτήριο ασφαλείας για να διασφαλίσει ότι τα τουρκικά πυρηνικά εργοστάσια θα τηρούν τα αυστηρότερα των κριτηρίων αυτών ασφαλείας. Επίσης θέλω να τονίσω ότι αυτή τη στιγμή γειτονεύομαι ε, με ένα από τα πιο επικίνδυνα πυρηνικά εργοστάσια του κόσμου, το Μέτσα στην Αρμενία, το οποίο είναι περίπου 16 χιλιόμετρα μακριά από τα ανατολικά σύνορα της Τουρκίας και αυτό αποτελεί σοβαρότατο κίνδυνο όπως γνωρίζετε λόγω της απειρχιωμένης τεχνολογίας που χρησιμοποιεί και θα είμαστε ευτυχείς εάν αυτό το ε, πυρηνικό εργοστάσιο έπαβε το ταχύτερο δυνατό τη λειτουργία του. Καλώς κατάλαβα ότι από αυτά τα οποία μας είπατε, ότι τα, τα κίνητρα αυτών που είναι υπέρ της πυρηνικής ενέργειας είναι τα ίδια σε όλες τις χώρες. Και τα ίδια ακούμε και στη Γαλλία. Δεν έχουμε ιδίους πόρους, οι τιμές θα αυξηθούν, θα δημιουργούν θέσεις απασχόλησης. Κοιτάξτε, πρέπει να πούμε ότι η πιο ακριβή ενέργεια ε, είναι ε, από την πυρηνική ενέργεια παράγεται, από την εκμετάλλευση πυρηνικών εγκαταστάσεων. Τώρα γιατί οι Γερμανοί έχουν προχωρήσει σε διαφορετικά μέτρα προωθώντας ε, την αποδοτικότητα, την αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης της ενέργειας ε, και ε, προτείνοντας την εκμετάλλευση και εναλλακτικών πηγών, όλα αυτά δείχνουν ότι υπάρχει μια έλλειψη, θα έλεγα, φαντασίας εν πολλής από αυτούς που υποστηρίζουν τα επιχειρήματα της πυρηνικής ενέργειας και νομίζω ότι δεν πείθετε, όπως δεν πείσατε και την κυρία Άτιτσι, η οποία επανήλθε, αν δεν κάνω λάθος. Είστε μαζί μας, κυρία Άτιτσι. Ε, θα έχουμε το ίδιο θέμα, η διαμηνία θα διακόψει όσο διαρκεί η τηλεδιάσκεψη με την Τουρκία γιατί δεν ακούμε στην καμπίνα τον ήχο. bonheur, on vous écoute. Ah,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 we also have this, I mean, uh, this uh, license in Akkuyu was given in 76. Επαναλαμβάνουμε ότι κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, επαναλαμβάνουμε ότι κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης δεν μπορεί να υπάρξει διερμηνία γιατί δεν ακούγεται στις καμπίνες. And uh, this uh, fault that is talked um,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 the people's needs and demands. And it is obvious that the Turkish people wants much more renewable energies and energy efficiency for our future. Um, okay. Merci beaucoup. You're right. Ευχαριστώ. Μπορείτε, αν θέλετε, να συνεχίσετε να μας ακούσετε, αν μπορείτε και να επανέλθετε στη συζήτηση αργότερα. Δεν ξέρω αν ακούσατε την αρχή της συνεδρίασής μας, της συζήτησής μας. Προφανώς δεν μας ακούτε, οπότε δεν θα μπορέσετε να επανέλθετε. Καλώς. Λοιπόν, αυτά ακούστηκαν κάποια επιχειρήματα. Ακούστηκαν λοιπόν κάποια επιχειρήματα και από την κοινωνία των πολιτών στην Τουρκία που αντιτίθεται στην οικοδόμηση μιας τέτοιας πυρηνικής μονάδας. Μας είπαν ότι τα επιστημονικά στοιχεία είναι αντιφατικά. Υπάρχει τεράστιο δυναμικό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, το οποίο δεν γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης και όλα αυτά έρχονται στους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τώρα για να μας πούνε τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις απαιτήσει της ενεργειακής πολιτικής, της ασφάλειας της πυρηνικής και τι ρόλο παίζουν τα θέματα αυτά στον τομέα των διαπραγματεύσεων με την Τουρκία, αν και γνωρίζουμε ότι το κεφάλαιο για την ενέργεια είναι κλειστό προς το παρόν και πρέπει η Τουρκία να αποδείξει ότι πράγματι είναι αποτελεσματική στον τομέα της ενέργειας. Λοιπόν, τι προϋποθέσεις υπάρχουν τι γίνεται με τις απαιτήσει σχετικά με τη μεταφορά του κοινοτικού κεκτημένου και ποια είναι η συζήτηση γενικότερα με την Τουρκία στον τομέα της ενέργειας. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Wolfgang Kilb Merci beaucoup, Madame la Présidente. Still the, little PowerPoint missing. Ε, περιμένουμε να αρχίσει η προβολή. Λέγομαι Wolfgang Kilp και είμαι ε, δικηγόρος στο Λουξεμβούργο σε θέματα πυρηνικής ενέργειας. Χαίρομαι που μου δίνετε την ευκαιρία να σας ε, μιλήσω και να κάνω μια σύντομη παρουσίαση επινομικών θεμάτων και υπόσχομαι να μην δείξω 397 διαφάνειες, να σας δηλητηριάσω. 27 διαφάνειες θα σας δείξω γρήγορα για να μην ε, πλήξετε από τις νομικές λεπτομέρειες. Η συνθήκη Ευρατόμ ακόμα ισχύει, η νομοθεσία Ευρατόμ για την πυρηνική ασφάλεια, η κατάσταση των πραγμάτων, διεθνεί υποχρεώσεις που απορρέουν από εδώ και κάποια συμπεράσματα. Αυτή είναι η δομή της ομιλίας μου. Ε, συγγνώμη, είναι περιορισμένη η τεχνογνωσία μου στους ε, υπολογιστές. Αυτή πάντως είναι η νομική μας πυραμίδα με τη συνθήκη Ευρατόμ, ε, το σύνταγμά μας αν θέλετε, στην κορυφή το δεσμευτικό δίκαιο, η οδηγία για την πυρηνική ασφάλεια που είναι ο πυρήνας εδώ και μετά το μη δεσμευτικό δίκαιο όπως γνωμοδοτήσεις απόψεις. Ακόμα υφίσταται η συνθήκη Ευρατόμ και μοιράζεται θεσμικά όργανα προϋπολογισμό με τη συνθήκη της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη συνθήκη για τη λειτουργία της. Διατηρεί όμως ε, τι δικές της ε, νομοθετικές διαδικασίες. Ε, ως επιτοπλίστων το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, λυπάμαι που το λέω εδώ αυτό, δεν συναποφασίζει, αλλά γνωμοδοτεί. Ο μεγάλος πλανήτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ένα μικρό δορυφόρο που περιστρέφεται γύρω της και που είναι η Ευρατόμ, λοιπόν. Η συνθήκη της ε, Ευρατόμ είναι η παλιά συνθήκη που ουσιαστικά ποτέ δεν τροποποιήθηκε μετά το 1958. Πολλά ε, είναι τα αντικείμενά της και με κόκκινο ή πορτοκαλί έχω αναδείξει ε, θέματα που αφορούν την νομοθεσία μας σχετικά. Υγεία και ασφάλεια αποσκοπεί στην προστασία της υγείας των εργαζομένων και του κοινού από την ιοντίζουσα ακτινοβολία, ε, θέτει ε, ενιαία πρότυπα ασφαλείας και φροντίζει να εφαρμόζονται, παρακολουθεί το επίπεδο της ραδιενέργειας στην ατμόσφαιρα, στα ύδατα και στο έδαφος και είναι έτοιμη, εάν υπάρξει κάποιο πρόβλημα, να αντιδράσει σε κατεπίγουσες ανάγκες. Αυτό ε, ζητεί η συνθήκη ευρατόμου από τα κράτη-μέλη. Αυτό είναι ένας άλλος τρόπος ε, να παρουσιάσουμε την ομοθεσία, το προσπερνώ γρήγορα αυτό και εδώ βλέπουμε πόσο περίπλοκα, ε, περίπλοκο είναι το δευτερογενές δίκαιο. Υπάρχουν βασικά πρότυπα ασφαλείας που είναι η βάση και τομεακές οδηγίες και κανονισμοί έχουμε την οδηγία για την πυρηνική ασφάλεια που είναι πολύ σημαντική και που θα πρέπει μέχρι τις 22 Εβδόμου τρέχοντος έτους να μεταφερθεί στις εθνικές νομοθεσίες. Ε, αυτή είναι μια οδηγία που συζητείται τώρα, που είναι η οδηγία για τα πυρηνικά απόβλητα, που δεν αφορά την ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων καθ' αυτών, αλλά με το κληροδότημα που αφήνουν, τι αφήνουν ως απόβλητα ε, μετά από τη διαδικασία παραγωγής πυρηνικής ενέργειας. Ποιο είναι το κλειδί τώρα της οδηγίας για την ε, πυρηνική ασφάλεια. Ε, είναι ότι δίνει ένομο ισχύ δεσμευτική σε πρότυπα διεθνή για την ασφάλεια, όπως είναι της Διεθνούς Υπηρεσίας Πυρηνικής Ενέργειας και τη Σύμβαση Πυρηνικής Ενέργειας. Έτσι, για την ασφάλεια, την πυρηνική ασφάλεια έτσι μπορούν να εφαρμόζονται ε, υποχρεωτικά. Επίσης, ε, παγιώνει την εθνική ευθύνη της πυρηνικής ασφάλειας, για την πυρηνική ασφάλεια από τα κράτη-μέλη, ε, ενισχύει τον ρόλο την ανεξαρτησία και τα μέσα εθνική, των εθνικών κανονιστικών αρχών, ενισχύει την ευθύνη των κατοχών της άδεια και προάγει τη συνεχή βελτίωση ε, των εγκαταστάσεων και προτύπων και από άλλες χώρες, όπως η ε, Τουρκία, γιατί υπάρχουν και οι εξωτερικές σχέσεις. Η Ευρατόμ ε, ε έχει υπογράψει, τις, μετέχει στις διεθνείς συμβάσεις και θέλω να τονίσω ποια είναι η σχέση ε, μεταξύ αυτής, αυτών των συμβάσεων και της κατάστασης στην Τουρκία. Υπάρχει η Σύμβαση για την Πυρηνική Ασφάλεια που λέει ρητά και κάποιοι ε, βουλευτές ενδιαφέρονται για αυτό το θέμα. Προβλέπει λοιπόν ότι κάθε συμβαλόμενο μέρος ε, θα αξιολογήσει όλους τους παράγοντες που αφορούν την συγκεκριμένη περιοχή. Αυτό έγινε για το σεισμικό κίνδυνο από τον καθηγητή Γκουλκάν και η Κομισιόν προφανώς καλεί τον καθένα και τα κράτη-μέλη να εξετάσουν το θέμα της επιλογής της περιοχής για οποιαδήποτε πυρηνική εγκατάσταση ως προς το σεισμολογικό κίνδυνο. Και έχει υπογράψει τη σύμβαση αυτή και η Τουρκία και η Ευρατόμ. Οπότε αυτό ε, έχει ε, κλείσει ως κεφάλαιο, είναι βέβαιο. Υπάρχει και μια άλλη σύμβαση που αφορά τα αναλωμένα καύσιμα και τα ραδιενεργά απόβλητα, που επίσης προβλέπει ως υποχρέωση τον έλεγχο της περιοχής και η Κομισιόν καλεί την Τουρκία να ε, υπογράψει και αυτή τη σύμβαση και να ξαναεξετάσει το θέμα της επιλογής του τόπου, της περιοχής. Τώρα, για τους γείτονες, ε, οι συνάδελφοι από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Βουλγαρία ε, Προφανώ ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για αυτή την πτυχή. Η Σύμβαση για την Πυρηνική Ασφάλεια προβλέπει επίση ότι κάθε συμβαλόμενο μέρο ε, θα ε, διεξαγεί διαβουλεύσει με συμβαλόμενα μέρη στην γειτονική περιοχή τη προτινόμενη πυρηνική εγκατάσταση. Άρα λοιπόν η πρόσκληση είναι παρακαλώ να λάβετε υπόψη σα του γείτονε και να διαβουλευτείτε με αυτούς. Εμπροκειμένου για τα κουγιού έχουμε την Ελλάδα, την Κύπρο, για τη Συνόπη επίση υπάρχουν οι και βέβαια η τρίτη τοποθεσία ακόμα δεν υφίσταται. Το ίδιο ισχύει αν υπήρχε εγκατάσταση επεξεργασίας απορριμμάτων. Να διαβουλευτείτε με τους γείτονες εάν πρόκειται να κάνετε κάποιο από αυτά τα βήματα που προβλέπει η σύμβαση. Και επίσης υπάρχει και μια, ε, η σύμβαση ESPOD που είναι η Γενική Περιβαλλοντική Σύμβαση η οποία επίσης προβλέπει την ίδια υποχρέωση. Ενημερώστε τους γείτονες το ταχύτερο δυνατόν όταν σχεδιάζεται ε, οποιαδήποτε από αυτές τις εγκαταστάσεις. Και πάλι λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί την τουρκική δημοκρατία να ε, συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία και να ενημερώνει τους γείτονες επί όλων των δραστηριοτήτων. Τώρα, ε, ετοιμότητα, ε, ε προ, έγκαιρη ε, κοινοποίηση μετά από πυρηνικό ατύχημα, αυτό έγινε μετά το Τσερνομπίλ, καλούνται τα μέλη να συνάψουν ε, συμφωνίες διμερείς ή πολυμερείς μεταξύ κοντινών γειτονικών χωρών. Εάν κάποια μέρη η Τουρκία γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ίσως δεν είναι τόσο χρήσιμο να έχει διμερή συμφωνία με την Ισλανδία, εν προκειμένου, αλλά με τους πραγματικούς γείτονες. Και επίσης καλούμε την Τουρκία να σκεφτεί, να συνάψει τέτοιου είδους συμφωνίες, διμερείς συμφωνίες κοινοποίησης. Ίσως έχετε δει την αναφορά τη χθεσινή στον τύπο τα κριτήρια για το stress test ε, υπάρχουν, θα ισχύσουν από την 1η Ιουνίου και κάποιες γειτονικές χώρες της Ένωσης όπως Ελβετία, η Ρωσική Ομοσπονδία, Ουκρανία, Αρμενία καλούνται να συμμετέχουν επίσης σε αυτά τα stress test και ίσως και η Τουρκία θα θελήσει σε βάση προαιρετική θελοντική να συμμετέχει για τα δικά της εργοστάσια. με δύο λόγια. Προσέλθετε σε αυτές και ε, ε, υπογράψτε τις συμβάσεις αυτές αν δεν τις έχετε υπογράψει ε, για την πυρηνική ασφάλεια. Προσοχή στον τόπο επιλογής, ενημέρωση των γειτόνων σχετικά με τα σχέδια που υπάρχουν. Να σκεφτείτε ενδεχομένως το ενδεχόμενο σύναψης διμερών συμφωνιών. Να σκεφτείτε αν μπορείτε να συμμετέχετε στα stress test και να είστε έτοιμοι να εφαρμόσετε το δεσμευτικό δευτερογενές δίκαιο, ε, για παράδειγμα την οδηγία για την πυρηνική ασφάλεια. Αν στο μέλλον κάποια στιγμή προσχωρήσει η Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα υπάρχουν συγκεκριμένα καθήκοντα, όπως για όλα τα κράτη-μέλη, να κοινοποιείται η νομοθεσία ε, πριν από την εφαρμογή της. Θα πρέπει να υποβάλλονται σχέδια για οποιαδήποτε ε, διαχείριση απορριμμάτων, αποκομιδή, προγράμματα επενδυτικά, επίσης πρέπει να κοινοποιούνται, όπως και οι διεθνείς συμφωνίες. Όλα αυτά ε, τα μελετά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αποφαίνεται και γνωμοδοτή. Επίσης υπάρχουν και διασφαλίσεις. Υπάρχουν 150 συνάδελφοι που ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο και επισκέπτονται τα πυρηνικά εργοστάσια για να δουν πώς αντιμετωπίζονται ουράνιο, πλουτόνιο και εδώ υπάρχει ένα καθεστώς μοναδικό θα έλεγα διότι προβλέπει ε, εφαρμοστές ε, υποχρεωτικά ε, διατάξεις ε, απέναντι στις επιχειρήσεις και αυτό είναι το ίδιο άρθρο όπως και στη Συνθήκη Λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι το βασικό καθήκον όλων των κρατών μελών να συνεργάζονται. Πρέπει να διασφαλίζεται ότι πληρούνται υποχρεώσεις με βάση τη συνθήκη, δηλαδή η διευκόλυνση της επίτευξης των κοινοτικών στόχων και αποχή από οποιαδήποτε μέτρα που μπορούν ενδεχομένως να υπονομεύσουν την επίτευξη αυτών των στόχων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τις εξηγήσεις σας για ένα σαφέστατο θέμα. Αυτή είναι η δουλειά που έχει η Τουρκία μπροστά της, αν επιλέξει την ατυχή επιλογή της πυρηνικής ενέργειας. Προσπάθησα να το πω προσεκτικά. Ο κύριος Λουσιάν Σεσίλ από τη Γενική Διεύθυνση Διεύρυνσης τώρα έχει ενδιαφέρον pourront aborder discuter négocier avec les autorités turques. il suffit d'appuyer sur le bouton normalement. Voilà. Θα μας πει και τι γίνεται με τις διαπραγματεύσεις. Σε Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πράγματι ασχολούμαι με τα της πυρηνικής ενέργειας στη Γενική Διεύθυνση Διεύρυνσης εδώ και αρκετό καιρό. Στο παρελθόν είχαμε να ασχοληθούμε κυρίως με τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης μέσω του προγράμματος Φάρος για την πυρηνική ασφάλεια. Τώρα έχουμε ένα νέο μέσο το οποίο διεδέχθη το Φάρο που λέγεται ΙΠΑ, ε, μέσο για την προένταξη ουσιαστικά. Σχετικά με τη χρήση του συγκεκριμένου μέσου, και στον πυρηνικό τομέα στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τις υποψήφιες ή δυνητικά υποψήφιες χώρες να είναι συμβατές ε, με το κοινοτικό κεκτημένο. Γι' αυτό βοηθάμε λοιπόν τις ε, επιλέξιμες για το ΙΠΑ χώρες μέσω συγκεκριμένων προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας κυρίως, που απευθύνονται κυρίως προς τις υπηρεσίες πυρηνικής ασφάλειας, τις οποίες θέλουμε να έλθουν στο ίδιο επίπεδο με τις ομόλογες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, παρέχουμε επίσης και εξοπλισμούς όπου αυτό χρειάζεται. Κάνουμε κάθε προσπάθεια έτσι ώστε σε επίπεδο ραδιοπροστασίας και πυρηνικής ασφάλειας να βοηθήσουμε. Η ραδιοασφάλεια φυσικά είναι βασικό ε, τμήμα του κοινοτικού κεκτημένου και πρέπει να παρέχεται στο ίδιο επίπεδο με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξεκινήσαμε το πρόγραμμα ΕΙΠΑ το 2007 λοιπόν. Δυστυχώς όμως το πρόγραμμα αυτό δεν εφαρμόζεται στην Τουρκία λόγω της άρνησης της Τουρκίας να πάρει μέρος. Αρνείται η Τουρκία να πάρει μέρος. Εξεπλάγημεν από αυτό. Οι πρώτες επαφές ξεκίνησαν το 2005 με την Τουρκία όταν ανακηρύχθηκε υποψηφία χώρα. Προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε τη χώρα αυτή να τύχει των θετικών σημείων του προγράμματος Φάρος. Πήγαμε επί τόπου, συζητήσαμε με τους Τούρκους αρμοδίους στην πυρηνική ενέργεια, Ήμασταν έτοιμοι να χρηματοδοτήσουμε μια σειρά ολόκληρη προγραμμάτων προχωρήσαμε στην προετοιμασία των προγραμμάτων και κάποια στιγμή υπήρξε από την τουρκική πλευρά ένα βέτο. Όταν ξεκινήσαμε το πρόγραμμα ΙΠΑ, προτείναμε επίσης τους Τούρκους εταίρους να πάρουν μέρος στο πρόγραμμα αυτό. Βάλαμε μάλιστα στην άκρη ένα κάποιο ποσό για τη χρηματοδότηση του προγράμματος στην Τουρκία, αλλά εξακολουθούν να αρνούνται συστηματικά τη συμμετοχή τους. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κανένα πρόγραμμα επιτόπου, δεν είναι δυνατόν να έχουμε μια ξεκάθαρη άποψη για το τι ακριβώς γίνεται με το κοινοτικό κεκτημένο και τι όχι. Δεν έχουμε επαφή ουσιαστικά. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο ανασφάλειας και θέλουμε στο μέλλον τα πράγματα να βελτιωθούν γιατί εμείς εξακολουθούμε να είμαστε ανοιχτοί για την τουρκική συμμετοχή στα προγράμματά μας παροχής τεχνικής βοήθειας. Τίποτα άλλο. Έχουν ζητήσει όλοι οι συνάδελφοι τον λόγο, θα τους τον δώσω με πάρα πολύ μεγάλη ε, χαρά. Εδώ όμως κύριε Γκιούνερ Άλπ υπάρχει ένα ερώτημα. Η Τουρκία αρνείται κατηγορηματικά να πάρει μέρος στα προγράμματα για την πυρηνική ασφάλεια και την προστασία από τη ραδιομόλυνση. Γιατί. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τους φίλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις εξηγήσεις τους, λέει ο κύριος Γκιούνερ Άλπ. Παρατηρώ ότι ο διάλογος στον συγκεκριμένο τομέα δεν είναι σε ικανοποιητική κατάσταση. Αυτό οφείλεται στο ότι οι διαπραγματεύσεις ένταξης επί του κεφαλαίου 15 ενέργεια έχουν μπλοκάρει, έχουν παγώσει. Όπως ξέρουμε οι διαπραγματεύσεις αυτές έχουν παγώσει για πολιτικούς λόγους, κάτι το οποίο δεν έχει καμία σχέση με το θέμα το οποίο συζητάμε. Το Κοινοβούλιο επανειλημμένα άλλωστε έχει απευθύνει εκκλήσεις ε, μέσω των εκθέσεών του έτσι ώστε οι διαπραγματεύσεις αυτές να ε, ε, επανέλθουν σε λειτουργία. Αυτό εξηγεί την κατάσταση των επαφών σήμερα. Υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη τα οποία παγώνουν το άνοιγμα του κεφαλαίου αυτού. Ένα κεφάλαιο που αφορά ιδιαίτερα τις χώρες αυτές θα έλεγα. όταν υπάρξει άρση των αντιρρήσεων οι οποίες υπάρχουν από συγκεκριμένη χώρα γύρω από το θέμα αυτό, νομίζω ότι θα υπάρξει δυνατότητα περαιτέρω συνεργασίας με τις υπηρεσίες της Ένωσης. Ο κύριος Κουμουτσάκος. Θα πρέπει να φύγει ο κύριος Κουμουτσάκος γιατί έχει μια ε, σημαντική συνάντηση αρκετά μακριά από το... Η συζήτηση εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Και όχι μόνο ενδιαφέρουσα, πολύ χρήσιμη γιατί υπήρχαν πολλά νέα στοιχεία τα οποία κανείς πρέπει να λάβει υπόψη του όταν προσεγγίζει το θέμα που συζητάμε σήμερα. Εγώ έχω να κάνω ε, μία παρατήρηση και μία ερώτηση. Η παρατήρηση αφορά στην μόλις ε, τελευταία παρέμβαση του ε, Τούρκο Μονίμου Αντιπροσώπου. Πράγματι υπάρχουν κεφάλαια τα οποία είναι κλειστά. Ένα από αυτά είναι το κεφάλαιο ενέργεια αλλά αυτό δεν πιστεύω ότι είναι επαρκής λόγος ή επαρκής δικαιολογία για να μην γίνονται οι απαραίτητες κινήσεις προεργασίας και προετοιμασίας όπως αυτή στην οποία αναφέρθηκε ο εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης ε, της Επιτροπής πριν λίγο εν ώψη του γεγονότος ότι η ενταξιακή διαδικασία έχει προοπτική και βάθος χρόνου. Επομένως η προετοιμασία, η επικοινωνία και η πρόοδος ορισμένων ε, προγραμμάτων όπως αυτά στα οποία αναφέρθηκε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής δεν αντιβαίνουν τη λογική της, ε, δεν, δεν αντιβαίνουν στη λογική ότι πρέπει να προετοιμαστεί ένα κεφάλαιο το οποίο κάποια στιγμή όλοι ελπίζουμε ότι θα συμπληρωθούν οι προϋποθέσεις για να ανοίξει. Επομένως ε, δεν θα πρέπει ορισμένα πράγματα περισσότερο να προβάλλονται ε, ως δικαιολογίες παρά ως πραγματική πολιτική βούληση. Ε, η ερώτησή μου είναι μία και απλή και είναι προς όλους και ε, πάντως προς ε, και προς τον κύριο καθηγητή αλλά και προς την τουρκική πλευρά που είπε ότι είναι απολύτως ασφαλής η περιοχή, μπορούμε να προχωρήσουμε. Εγώ δεν έχω τις δυνατότητες και πιστεύω πολύ λίγοι από εμάς αυτήν την έχουν τις τεχνικές ή επιστημονικές δυνατότητες να κρίνουν σε βάθος το ζήτημα αυτό. Ένα όμως είναι βέβαιο ότι υπάρχουν υψηλές και ισχυρές αμφιβολίες για την καταλληλότητα, για την καταλληλότητα αυτής της περιοχής, η οποία είναι μια σεισμική περιοχή. Το γεγονός αυτό και μόνο ότι υπάρχουν υψηλές και θεμελιωμένες αμφιβολίες, ακόμα και στον τοπικό πληθυσμό, στην τοπική κοινή γνώμη, αλλά και ευρύτερα, θα έπρεπε να είναι ένας παράγων ανασταλτικός, πιστεύω, για την υλοποίηση του σχεδίου. Και επίσης δεν μπορώ παρά να ζητήσω κάποια διευκρίνηση σε αυτό που είπε η εκπρόσωπος της ε, Greenpeace σε σχετικά με την δανειοδότηση, το χρόνο δανειοδότησης και έγκρισης εγκατάστασης του, ε, του πυρηνικού εργοστασίου που έγινε, αν θυμάμαι καλά, το 1976, με άλλες συνθήκες και κάτω από άλλες τεχνικές δυνατότητες και γνώσεις, ενώ από τότε έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια και δεν έχει ανανεωθεί η συγκεκριμένη άδεια εγκατάστασης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Κουμουτσάκο. Κύριο Χατζηγεωργίου. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρέπει να πω ότι και για μένα ήταν ε, πολύ ενδιαφέρουσε οι πληροφορίε που άκουσα και από τον κύριο καθηγητή αλλά και από τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Γενικής Διεύθυνσης. Ε, είμαι σίγουρος καταρχήν ότι ε, παρά τα εκατέρωθεν επιχειρήματα νομίζω ότι ε, δεν μπορούν να προσθεθούν καινούρια. Είναι γνωστά τα επιχειρήματα όσων εναντιώνονται στην πυρηνική ενέργεια, είτε αυτή είναι προς χρήση πολεμική, είτε αυτή είναι προς χρήση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και είναι γνωστά τα αντεπιχειρήματα. Και δεν νομίζω ότι σε αυτή την αίθουσα μπορούμε να προσθέσουμε πολλά πράγματα. Εγώ πιστεύω ότι αν θα επιτευχθεί ο στόχος της αποπυρηνικοποίησης πρώτα απ' όλα της Ευρώπης και συνακόλουθα της μη δημιουργίας νέων πυρηνικών σταθμών όπως την παρούσα περίπτωση στην Τουρκία, αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνον εάν ογκούται συνεχώς το αντιπυρηνικό κίνημα. Και όσον αφορά την Τουρκία, θα μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος της μη υλοποίηση αυτής της ιδέας, κυρίως εάν ο τουρκικός λαός ε, δείξει έντονη αντίθεση σε αυτή την κίνηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, επίσης σαν θεσμικός οργανισμός, έχει ουσιαστικό ρόλο να διαδραματίσει, ε, κυρίως προς την κατεύθυνση των επαφών, ε, της ανάπτυξης των εκατέρωθεν συναντήσεων έτσι ώστε οποιοδήποτε αποτέλεσμα βγει στο τέλος να είναι αποτέλεσμα συνένεσης και αποτέλεσμα διαβούλευσης και με τα γειτονικά κράτη όπως επιβάλλεται και από την συνθήκη στην οποία αναφέρθηκε ο κύριος Χίλπ. Έχει λεχθεί ότι οι συζητήσεις έχουν παγώσει ή δεν υπάρχουν επαφές μεταξύ Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης για το θέμα αυτό, διότι είναι κλειστό το κεφάλαιο της ενέργειας και θέλω να προσθέσω ένα ακόμα επιχείρημα, ένα ακόμα επιχείρημα στα, όσα, έχει πει ο κύριος Κουμουτσάκος. Αν έχω καταλάβει καλά, αυτού του τύπου διαβουλεύσεις γίνονται και με κράτη που δεν έχουν κάνει αίτηση ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ουκρανία, Αρμενία. Άρα, δεν έχει να κάνει τίποτε αυτό με το αν είναι ανοιχτό ή κλειστό το, το θέμα της ενέργειας. Αντίθετα, επειδή εσείς είστε σε διαδικασία ένταξης, έχετε δύο λόγους περισσότερους από τα κράτη στα οποία αναφέρθηκα για να έχετε αυτού του τύπου τις επαφές. Θέλω επίσης να πω το εξής. Εγώ δεν είμαι αισιόδοξο για το μέλλον της ανθρωπότητας συζητάμε, καταλαβαίνετε, ένα ζήτημα που μας υπερβαίνει. Δεν αφορά μόνο τον τουρκικό λαό, αφορά και τους γειτονικού λαούς, αφορά όλη την Ευρώπη. Συζητούμε τώρα επειδή γίνεται μια προσπάθεια εγκατάσταση πυρηνικό σταθμό στην Τουρκία. Αφορά όλη την ανθρωπότητα. Και δεν είμαι αισιόδοξο ότι η ανθρωπότητα δείχνει να κατανοεί ότι μέσα στη θύελα δεν θα βρεθεί ένα θεϊκό χέρι να μας σώσει δείχνουμε να νομίζουμε ότι την κρίσιμη ώρα όταν μας έρθει το μεγάλο ατύχημα που τώρα νομίζουμε ότι μπορεί να μας έρθει από σεισμό αλλά κανένας δεν ξέρει αν οι κλιματικές αλλαγές στις επόμενες δεκαετίες θα φέρουν νέου τύπου ε, θεομηνίες. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω ότι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ενισχύσουμε την πίστη του τουρκικού λαού στη συγκεκριμένη περίπτωση ότι πρέπει να σηκώσει ανάστημα και να εμποδίσει, ναι, ε, την τουρκική κυβέρνηση από το να προχωρήσει σε ένα εγχείρημα το οποίο εμπεριέχει, όλοι το έχουμε στο μυαλό μας, ακόμα και αυτοί που υποστηρίζουν ότι πρέπει να κάνουν πυρηνικό σταθμό, μέσα στο μυαλό τους υπάρχει ο φόβος. Υπάρχει πίσω από το μυαλό η σκέψη ότι μην την πατήσουμε κάποια στιγμή. Παρόλα αυτά ε, δεν παίρνουμε ε, την κρίσιμη απόφαση ε, υιοθέτηση της πιο σωστής ε, ιδέας. Εγώ θέλω να κλείσω με το εξής. Αναφερθήκαμε σε κινδύνους που μπορεί να προέρθουν από σεισμική δραστηριότητα και υπήρξαν οι απαντήσεις από τον κύριο καθηγητή υπήρξε η δική μου τοποθέτηση ότι αύριο μπορούμε να δούμε και νέου τύπου ε, κλιματικές αλλαγές που θα φέρουν άλλου τύπου θεομηνίες πέρα από τους σεισμούς ε, και τις ε, ε οποιασδήποτε άλλες ε, θεομηνίες γνωρίζομαι. Αλλά ήθελα να ρωτήσω, είμαστε βέβαιοι ότι οι πυρηνικοί σταθμοί δεν εμπεριέχουν ένα μεγάλο κίνδυνο από τυχόν τρομοκρατική επίθεση. Αυτό βλέπω ότι δεν υπάρχει καν στις συζητήσεις που γίνονται ε, για την κατάργηση της ε, παραγωγής ε, ηλεκτρισμού από πυρηνική ενέργεια, ενώ την ίδια ώρα βλέπουμε ότι το τρομοκρατικό κίνημα παγκόσμια έχει τα τελευταία χρόνια δείξει τα, τα δόντια του. Ε, όσον αφορά τα ωφέλη, τα οικονομικά, θα πω μόνο το εξή. Η Ιαπωνία είχε ωφέλη οικονομικά από αυτό το πράγμα για πάρα πολλέ ε, δεκαετίε. Τα έχασε μέσα στου τελευταίου έξι μήνε. Αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Merci beaucoup, Madame Keller, Κυρία Keller, μετά κυρία Θεοχάρους, μετά κυρία Παπαδοπούλου. Μιλάμε πολύ για πυρηνικές απειλέ, τρομοκρατικέ ε, ε Τα νέα κράτη-μέλη πολλέ φορές αρνούνται να εξετάσουν, να κάνουν δοκιμές ε, στα εργοστάσια ε, απέναντι σε ε, ενδεχόμενα πυρηνικά τρομοκρατικά πλήγματα ή συντριβή αεροσκαφών που μπορεί να είναι ένα πιο ευρύ πρόβλημα. Υπάρχουν λοιπόν όλα αυτά τα προβλήματα. Επιλογή της τοποθεσίας του πυρηνικού εργοστασίου είναι ένα πρόβλημα αυτό και στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί υπάρχουν πυρηνικά εργοστάσια τα οποία βρίσκονται πάνω σε γραμμή ρήγματος και ήθιστε τα πυρηνικά εργοστάσια ή τα σημεία αποκομιδής των πυρηνικών αποβλήτων να γίνονται στα σύνορα με άλλες χώρες. Αυτό γίνεται και το βλέπουμε πολλές, σε πολλά σημεία των σύνορων. Μπορεί να υπάρχουν πολλές απειλές ε, από ατυχημάτων, από σεισμό, λόγω της αλλαγής του κλίματος κλπ. Ε, δύσκολα ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος, γιατί είναι πολύ κίνδυνοι. Επίσης, ερωτήσεις σχετικά με κινδύνους που μπορεί να ακούγονται ανόητοι, αλλά αυτό που μας λένε συνήθως είναι τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα τουρκικά πυρηνικά εργοστάσια. Αν δω πόσα λίγα μπορούμε να κάνουμε για τα πυρηνικά εργοστάσια στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, αναρωτιέμαι πώς θα βελτιώσουμε την κατάσταση εκτός Ένωσης. Τι ερώτηση, τι μπορείτε εσείς να κάνετε και στο έδαφος της Ένωσης και εκτός Ένωσης για τα πυρηνικά εργοστάσια. Μπορούμε να κάνουμε τίποτα, μπορούμε να επηρεάσουμε το πού θα εγκατασταθούν, πού θα κατασκευαστούν, να ε, καταδείξουμε κινδύνους ασφαλείας. Τι μπορούμε να κάνουμε. Μιλήσατε για μια νομική βάση στις συνθήκες που λέει ότι θα πρέπει να εξετάσετε την ε, επιλογή τοποθεσίας. Πολλά μπορεί να εξετάσετε, αλλά τι βγαίνει. Και βέβαια ε, οι γείτονε ε, τους οποίους διαβολεύονται δεν είναι κράτη-μέλη. Άρα λοιπόν ποια είναι η απάντηση που θα δοθεί στον πολίτη ο οποίος ρωτάει και ζητάει να μάθει τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και για τα πυρηνικά εργοστάσια στην Τουρκία αλλά και για τα πυρηνικά εργοστάσια στο έδαφος τη Ένωση. Τώρα, αν προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει η Τουρκία να προσχωρήσει και στη συνθήκη Ευρατόμ, υποθέτω, έτσι δεν είναι. Μάλιστα, αυτό μου το απαντήσατε απευθεία. Καλώ ευχαριστώ. Αυτά είχα να ρωτήσω. Ευχαριστώ, κυρία Κέλλερ. Κυρία Θεοχάρου. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Βρίσκομαι εδώ όχι μόνο ως βουλευτής της Κυπριακής Δημοκρατίας, μιας χώρας που απέχει μόνο 40 χιλιόμετρα από το IQU, αλλά και ως μέλος οικολογικών οργανώσεων σε όλο τον κόσμο που αγωνίζομαι εναντίον των πυρηνικών και των εργοστασίων και της πολεμικής χρήσης, αλλά και ως γιατρός που έχω ασχοληθεί με θύματα του Μετζαμόρ, του Σέμι Παλάτινσκ, του Τσέρνομπιλ για πάρα πολλά χρόνια. Συνεπώς, η έγνοια μου δεν αφορά ειδικά μόνο την Τουρκία, παρόλο που είναι τόσο πολύ κοντά στο νησί μου, που θα έλεγε κάποιος ότι... Αλλά μια πυρηνική απειλή μπορεί να πλήξει ολόκληρη την Ευρώπη και συνεπώς τα μέτρα πρέπει να αφορούν ολόκληρη την Ευρώπη. Ναι, βλέπω αυτή τη στιγμή το πρόβλημα με την Τουρκία, αλλά δεν θέλω να επιβάλλουμε αυστηρότερους όρους για την Τουρκία. Πρέπει η Τουρκία να συμμορφωθεί με τα διεθνή θεσμία και πρέπει όσοι δεν συμμορφώνονται να έχουν την ανάλογη τιμωρία. Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι τα εξή. Ο καθηγητή Γκιουλκάν μα είπε ότι οι πιο κατάλληλε περιοχέ είναι η Συνόπη και το Άκυγιου. Ωστόσο υπάρχει η μελέτη στην οποία αναφερθήκατε του Westaway που λέει ότι είναι πέρα για πέρα επικίνδυνη και καταστροφική η εγκατάσταση σε αυτά τα εργοστάσια. Πώς μπορούν να συμβιβαστούν αυτά τα δύο. Το δεύτερο, ο τουρκικός λαός έχει ενημερωθεί επαρκώς και ποια είναι η αντίδραση του τουρκικού λαού σε αυτό τον κίνδυνο. Το τρίτο ερώτημα αφορά βέβαια τον εξοχότατο πρέσβη, τον κύριο Γκιουνεράλπ. Ε, έχετε διαβουλευθεί με την Κυπριακή Δημοκρατία και τα άλλα κράτη που πιθανόν να, ενημερω... να υποστούν τις συνέπειες εύχομαι ποτέ να μην συμβεί αλλά αν συμβεί κάποιο πυρηνικό ατύχημα όπως προνοούν και οι συνθήκες που αναφέρθηκαν. Και το τέταρτο εξοχότατε έχει μήπως μπορείτε να διαψεύσετε τη δήλωση του κυρίου Νταβούτογλου, του Υπουργού Εξωτερικών της χώρας σας, ότι αν η Κύπρος, η φτωχή η μικρή Κύπρος, προχωρήσει σε εκμετάλλευση των αποθεμάτων υδρογονανθράκων που έχει στην αποκλειστική οικονομική της ζώνη, αυτό θα είναι αιτία πολέμου για την Τουρκία. Σας ευχαριστώ. Merci, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Έχω παρακολουθήσει με πολύ ενδιαφέρον όλες τις συζητήσεις και ιδιαίτερα τις δύο τελευταίες ε, για το νομικό πλαίσιο αλλά και επίσης για τη θέση της Κομισιόν και με φοβίζει πραγματικά το γεγονός ότι ε, η Τουρκία δεν έχει υπογράψει συμβάσεις, ότι όπως έχει αναφερθεί από τον ε, κύριο Κίλπ, πρέπει προτού σχεδιαστούν τέτοιες εγκαταστάσεις να υπάρχει ενημέρωση των γειτόνων και μιλά για τους πραγματικούς γείτονες. Η χώρα μου, η Κύπρος, είναι πραγματικός γείτονας, γιατί όπως έχει πει και η κυρία Θεοχάρους, είναι μόνο 40 χιλιόμετρα μακριά αλλά είναι χώρα ευρωπαϊκή. Επομένως, οι ανησυχίες της Ευρωπαϊκής Κύπρου είναι και ανησυχίες ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Τουρκία δεν έχει κοινοποιήσει την πρόθεση της για να δημιουργήσει αυτόν τον πυρηνικό σταθμό, είτε στη Σινόπιν είτε στο ΑΚΙου. Και εμείς πραγματικά μας ενδιαφέρει το γεγονός ότι έτσι τελικά έχει προχωρήσει με συμφωνία με τη Ρωσία και μάλιστα θα είναι έτοιμος αυτός ο πυρηνικός σταθμός το 2020. Επομένως, εμείς συζητούμε, έχοντας ως δεδομένο, ότι η Τουρκία αποφάσισε, υλοποιεί, έχει σχεδιάσει ερήμην των γειτόνων της. Επομένως, το πρώτο μου ερώτημα είναι τι μπορεί να γίνει τώρα, διότι μιλούμε εκ των υστέρων. Η Τουρκία αποφάσισε, υλοποιεί. Δεύτερη ερώτηση. Άκουσα την ακτιβίστρια ε, από την Τουρκία που μιλούσε για την έλλειψη διάλογου με τον τουρκικό λαό. Και κοιτάζοντα τι σημειώσει που έχουμε ενώπιον μα, φαίνεται ότι ένα σημαντικό ποσοστό, πέραν του 80% των κατοίκων τη Μεσίνα, τη περιοχή του Άκιου, των περιοχών που γειτονιάζουν με τη Μεσόγειο, είναι σφόδρα εναντίον τη εγκατάσταση πυρηνικών σταθμών, γιατί ακριβώ η περιοχή του Άκιου είναι σεισμογενή. Βρίσκεται 25 χιλιόμετρα μόνον από σεισμογενή γραμμή ρήγματος. Και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Επομένως, γιατί οι τουρκικές αρχές δεν ακούν τη φωνή του τουρκικού λαού. Εάν δεν ακούν τον τουρκικό λαό, πόσο μάλλον να ακούσουν εμάς τους γείτονες που δεν είμαστε νηπικοί της Τουρκίας. Αυτή είναι η δεύτερη με ερώτηση. Η τρίτη ερώτηση. Θα συμφωνήσω, κυρία Φλότ, μαζί σας απόλυτα, όταν έχετε πει ότι υπάρχει έλλειψη φαντασίας Είμαι χημικό στο επάγγελμα και για πολλά χρόνια παρακολουθώ το θέμα των πυρηνικών. Μάλιστα συμμετείχα ενεργά σε παρόμοιε συζητήσει στο Συμβούλιο τη Ευρώπη για 9 συναπτά έτη. Η πυρηνική ενέργεια και η πυρηνική σταθμή δεν είναι η λύση. Η λύση σήμερα για προστασία του περιβάλλοντο, για ασφάλεια του πλανήτη μα και δεν μιλούμε μόνο για την Κύπρο ή για την Τουρκία ή για την Ευρώπη, μιλούμε για τον πλανήτη ολόκληρο πρέπει να μας προωθήσει να βρούμε υπαλλακτικές λύσεις. Και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι μια λύση. Γιατί να προσφύγουμε σε, πυρηνικά, ε, σε πυρηνικούς αντιδραστήρες και πυρηνικά εργοστάσια. Τι άλλες υπαλλακτικές επιλογές είχαν η Τουρκία και οι αρμόδιες τουρκικές αρχές. Εξετάστηκαν. Τι έρευνε έγιναν, γιατί ευρέθηκε ότι η μοναδική λύση κλειδί είναι το ο πυρηνικό αντιδραστήρα. Εγώ θα ήθελα να δω μελέτε αν εξετάστηκαν άλλε συμπαλλακτικέ λύσει και αν έχετε τέτοιε συμπαλλακτικέ, δώστε μα εδώ έναν executive summary το οποίο να μελετήσουμε. Και η τελευταία μου ερώτηση αφορά ακριβώ αυτά τα υπονοούμενα που άφησε ο κύριο Πρέσβη εδώ, ότι κάποιε χώρε αντιτίθενται όσον αφορά το άνοιγμα κεφαλαίου για την Τουρκία. Αυτό, αγαπητή κυρία Φλότ, το ακούμε εδώ και δύο χρόνια. Είμαστε νέοι ευρωβουλευτές από την Κύπρο, γιατί η χώρα μας ευτυχώς εντάχθηκε το 2004 στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τολμώ να πω ότι η Τουρκία έχει το κλειδί αν θέλει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτον και κύριον έχει προσυπογράψει πρωτόκολλα, όπως το πρωτόκολλο της Άγκυρας. Δεν το έχει υλοποιήσει. Ας το υλοποιήσει. Η Κύπρος δεν άσκησε βέτο εναντίον της ενταξιακής πορείας της Τουρκίας, αλλά ζητά το αυτονόητο να μπορεί η Τουρκία ό,τι υπογράφει να το εφαρμόζει. Και ερώτηση μου είναι στον κύριο Κίλπ. Κύριε Κίλπ, εμεί έχουμε την εμπειρία να έχουμε μια γείτονα χώρα, την Τουρκία, που κατέχει 37% των εδαφών μα και δυστυχώ ό,τι υπογράφει δεν το υλοποιεί. Πώ εσεί μπορεί να είστε βέβαιο ότι χωρί να μπει στην Ευρώπη ή όταν μπει στην Ευρώπη θα εφαρμόσει όλα αυτά τα οποία νομικά θα πρέπει να την δεσμεύσουν. Προσωπικά αφισβητώ αν à το πράξει. Euh, λοιπόν, επανερχόμεθα εδώ σε αυτούς που πήραν το λόγο. Δεν ξέρω αν και η κυρία Τίτσι επανέλθει με την τηλεδιάσκεψη. Λοιπόν, το κεφάλαιο δεν έχει παγώσει σε επίπεδο α, σε επίπεδο θα έλεγα αντιστάθμισης του παγώματος του πρωτοκόλου της Άγκυρας, έτσι δεν είναι. Είναι τμήμα των κεφαλαίων τα οποία έχουν, δεν έχουν ανοίξει είτε από τη Γαλλία είτε από την Κύπρο, αλλά δεν είναι σαν κύρωση για, το μη, ε, για τη μη ε, υπογραφή, για το μη σεβασμό μάλλον του πρωτοκόλου της Άγκυρας. Κυρία Άτιτσι, είστε μαζί μας, ακούσατε τη συζήτηση. Επανερχόμεθα σε εσά λοιπόν. Διακόπτουμε πάλι την διευμηνία. Εγώ δεν άκουσα, λέει χοντρικά η κυρία από την Τουρκία, τι είπαν οι Έλληνες συνάδελφοι, γιατί δεν έχω μετάφραση εδώ, δεν ακούμε. Γενικά η διερμηνία δεν μπορεί να λειτουργήσει στα πλαίσια του Skype. Δεν λειτουργεί η διερμηνία στα πλαίσια του Skype. Euh, α, κοιτάξτε, νόμιζα ότι κάποιοι από τους βουλευτές που μίλησαν αναφέρθηκαν και στα δικά σας επιχειρήματα σχετικά με την αντίθεση του πληθυσμού, ιδιαίτερα αυτών οι οποίοι είναι κοντά στις προβλεπόμενες εγκαταστάσεις. Στην ουσία υπήρχε μια επανάληψη των δικών σας περισσότερων επιχειρημάτων. Θα ήθελα να μάθω πώς προβλέπονται οι συνέχειες των κινητοποιήσεων στην Τουρκία, στον τομέα της ενέργειας, του περιβάλλοντος, σε επίπεδο δημοκρατίας οι, οι κινητοποιήσεις αυτές έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Ποιες είναι οι προοπτικές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 Euh, euh, λοιπόν, ακούσατε ίσως θα πρέπει στην επόμενη συνάντησή μας ε, στην Τουρκία να συναντηθούμε με το δίκτυό σας, γιατί υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες και πολλές ενδιαφέρουσες συζητήσεις, οι οποίες ακούστηκαν, και θα επανέλθουμε όταν έλθουμε εν αντιπροσωπεία στην χώρα σας. Σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας, λέει η Πρόεδρος. Ο πρέσβης Κιούνερ Αλπ έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να πω ότι συμφωνώ με αυτά τα οποία είπατε προηγουμένως, μετά από την πρώτη παρέμβασή μου, ότι δηλαδή τα επιχειρήματα τα οποία εκφράζονται από τις δύο πλευρές υπέρ ή κατά της πυρηνικής ενέργειας είναι τα ίδια σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα στην Ευρώπη. Δεν είναι δηλαδή, εμεί στην Τουρκία δεν εφεύραμε την πυρίτιδα, ε, δεν ε, ανοίξαμε μια συζήτηση που δεν υπήρχε, τα επιχειρήματα και η συζήτηση είναι ανοιχτή. Το κόστος της ενέργειας και το θέμα της ύπαρξης άλλων ενεργειακών πόρων είναι θέματα τα οποία ε, ακούγονται παντού και στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την ιδιαίτερη κατάσταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Τουρκία είναι αλήθεια ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο δυναμικό ηλιακής αιωλικής επίσης αλλά όπως όλοι γνωρίζουμε είναι ενέργειες οι οποίες, μορφές ενέργειας οι οποίες κοστίζουν ιδιαίτερα και δεν μπορεί να επιβιώσουν αν δεν επιδοτούνται για τη βιοθερμία στην οποία αναφέρθηκε η κυρία Αλτιτζή, Ατιτσή μάλλον, έχουμε δυνατότητες μεγάλες, αλλά από ό,τι γνωρίζω δεν μπορεί η βιοθερμία να αποτελέσει παρά μόνο μια συνοδευτική πηγή ενέργειας. Η συζήτηση πάντως συνεχίζεται. Διαπιστώνω ότι σε περίοδο προεκλογικής εκστρατείας Ξέρετε ότι υπάρχουν εκλογές σε 15 μέρες στην Τουρκία. Διαπιστώνω λοιπόν ότι στα πλαίσια αυτού του κλίματος όπου όλα συζητιούνται το θέμα της ενέργειας δεν φαίνεται να απασχολεί τις πυρηνικές ενέργειες, δεν φαίνεται να απασχολεί ε, τον κόσμο. Ίσως γιατί όλα τα πολιτικά κόμματα τα οποία ε, είναι υποψήφια συνειδητοποιούν ότι τελικά ότι έχουν γίνει υπολογισμοί και δεν υπάρχει κάποιος λόγος περισσότερη συζήτηση σε αυτό το επίπεδο. Η χρήση λοιπόν της πυρηνικής ενέργειας δεν αμφισβητείται από τα μεγάλα πολιτικά κόμματα της χώρας μου. Αυτό είναι κάτι το οποίο οφείλω να υπογραμμίσω. Για τον κύριο Χατζηγεωργίου, αναφέρθηκε στη συνεργασία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κάποιες γειτονικές χώρες. Αυτό το οποίο προτάθηκε χτες είναι μια συνεργασία σε εθελοντική βάση, τα λεγόμενα stress test και με την Αρμενία και με την Ουκρανία επί τη βάση της έκκλησης που απευθύνεται από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τις χώρες αυτές σε, σε εθελοντική βάση. Δεν είναι νομικά δεσμευμένες οι χώρες αυτές. Δεσμευτικές προτάσεις μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μόνο προς τα κράτη-μέλη. Ίσως η εξήγηση αυτή να μην είναι ικανοποιητική για όλους, αλλά επαναλαμβάνω ότι το κεφάλαιο 15 δεν είναι υποσυζήτηση, δεν είναι ευθύνη της Τουρκίας αυτό, οπότε είναι πολύ λογικό για την Τουρκία να προχωρά σε μονομερή μέτρα θα έλεγα στον συγκεκριμένο τομέα. Για μια ακόμη φορά σωστά υπογραμμίσατε Πρόεδρε ότι το άνοιγμα του κεφαλαίου 15 έχει ε, μπλοκάρει, αν θέλετε, μονομερός από το Συμβούλιο από το 2006. Και για μια ακόμη φορά απευθύνω έκκληση στους φίλους της χώρας που μπλοκάρουν αυτή τη διαπραγμάτευση να ενθαρρύνουν την κυβέρνησή τους να οδηγηθεί σε μια αλλαγή θέσης. Η κυρία Θεοχάρους αναφέρθηκε στη διαχείριση των υδρογων ανθράκων γύρω από την Ίσο Κύπρο. Ε, η θέση της Τουρκίας είναι σαφής. Οι πόροι αυτοί ανήκουν και στις δύο κοινότητες και εφόσον δεν έχει υπάρξει συμφωνία για το μέλος της Κύπρου, της νήσου Κύπρου λέει ο μιλητής, τότε δεν θα ήταν νομίζω σωστό να ξεκινήσει κανείς την εκμετάλλευση, έστω και τη διαδικασία ανείχνευσης των συγκεκριμένων αυτών ενεργειακών πόρων. Είναι ξεκάθαρη θέση μας γύρω από αυτό. Δεν έχω νομίζω κάτι επιπλέον να προσθέσω, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την πρωτοβουλία που αναλάβατε. Καλώς. Υπήρξαν κάποιες ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την κατάσταση των σχέσεων και την εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου και τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να βοηθήσει την Τουρκία πιθανώς να διαμορφώσει μια ενεργειακή πολιτική χωρίς πολιτική ε, στον τομέα, χωρίς πυρηνική παρέμβαση. Σύντομα όμως, γιατί δεν έχουμε δυστυχώς χρόνο, έχουμε φτάσει στο, τέλος της συνεδρίας ουσιαστικά. Μπορώ να μιλήσω στα γερμανικά. Πολύ σύντομα ε, για τις ερωτήσεις της κυρίας Κέλλερ. Πρώτον, το άρθρο 194 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει ότι κάθε κράτος μέλος αποφασίζει για το ενεργειακό του μείγμα. Στην Ευρώπη 14 χώρες έχουν και 13 δεν έχουν πυρηνικά. Τώρα, για την ε, επιφυλακτικότητα ορισμένων γερμανόφωνων ε, χωρών απέναντι στην πυρηνική ενέργεια δεν θα σας μιλήσω. Τώρα, η βασική ευθύνη για την ε, ασφάλεια είναι στους υπεύθυνους για την επιχείρηση και τα κράτη-μέλη. Οι επιθεωρητές δεν εξετάζουν την ασφάλεια του πυρηνικού ε, εργοστασίου, ε, εξετάζει μόνο αν το θόριο, ουράνιο, ε, πλουτόνιο υπάρχουν στις δηλωθήσεις ποσότητες, δηλαδή είναι περιορισμένο το καθήκον των επιθεωρητών. Τρίτον, όπως είπε σωστά ο πρεσβευτής, τα τέστα αντοχής για μη κράτη-μέλη της Ένωσης αυτονοήτως ε, είναι δυνατά μόνο σε προαιρετική βάση. Δεν γίνεται άλλωστε και διαφορετικά. Τέταρτον, οι διεθνείς υποχρεώσεις της Τουρκίας, για παράδειγμα που απορρέουν από τη Σύμβαση για την Πυρηνική Ασφάλεια, μπορούν στην Ευρώπη μόνο τότε να ε, ισχύσουν και να επιβληθούν αφού η Τουρκία γίνει μέλος και άρα θα έχει ε, εφαρμογή η οδηγία για την πυρηνική ασφάλεια και στην Τουρκία. Αλλιώς είναι καθαρά διεθνής, ε, διεθνούς δικαίου η υπόθεση αυτή. Ευχαριστώ. Ο συνάδελφός σας από τη Γενική Διεύθυνση Διεύρυνσης έχει να προσθέσει κάτι ή ο καθηγητής. Ναι. Ε, ευχαριστώ. Ε, θα είμαι πολύ ευτυχής να αναφέρω και να τις ε, πολύ λεπτές ερωτήσεις που ετέθησαν στον κύριο Πρεσβευτή, γιατί αφορούν θέματα προσχώρησης μέλλοντος πολιτικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενδεχομένως της Τουρκίας. Εγώ θα ήθελα να απαντήσω στην κυρία Θεοχάρους, η οποία αναφέρθηκε στην ε, απόκληση των δηλώσεων μου, ότι δηλαδή αφενός είναι ασφαλής οι δύο τοποθεσίες και αφετέρου ότι υπάρχει πιθανή σεισμογενής δραστηριότητα και στις δύο αυτές περιοχές. Αν μου επιτρέπετε, κυρία Πρόεδρε, θα μιλήσω ως μηχανολόγος για το περιορισμένο αντικείμενό μου. Ως ε, τεχνολόγοι, η τεχνολογικοί ειδικοί, θέλουμε να υπηρετήσουμε τις κοινωνίες. Τι θέλουμε δηλαδή, να έχουν υγιείς εγκαταστάσεις, να έχουν μεταφορικά δίκτυα, να έχουν ό,τι άλλο συλλογικά χαρακτηρίζεται ως ε, ε, κοινωνία. Ε, τζάμπο αεροσκάφη, υψηλά κτίρια κλπ. Είναι το συλλογικό καθήκον των μηχανολόγων να εκτιμούν επί τη βάση εμπειρικών δεδομένων ή καμιά φορά και επί τη βάση θεωριών ποιες μπορεί να είναι οι εξωτερικές επιδράσεις για το προσκατασκευή έργο το ανθρωπογενές αυτό οικοδόμημα. Όταν πρόκειται για το σχεδιασμό ενός πυρηνικού εργοστασίου, εξετάζομαι με βάση τις ε, γνώσεις μας ποιες εξωγενείς επιδράσεις μπορεί να το επηρεάσουν μετά από κάποιο διάστημα, μετά την κατασκευή δηλαδή της εγκατάστασης. Τι θα το επηρεάσει και τι μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο έτσι για την κοινότητα και τη γειτονική περιοχή. Και ε, ο κίνδυνος δεν περιορίζεται βέβαια στα εθνικά σύνορα. Η απάντηση λοιπόν που θα σας δώσω εδώ είναι εξετάζομαι τη σεισμογενή δραστηριότητα στις δύο περιοχές και μετά κάνουμε ένα, κατασκευάζομαι ένα πιθανό σενάριο, όχι ακριβές βέβαια καθόλου, ε, λαμβάνοντας υπόψη κάποιο επίπεδο σεισμογενή δραστηριότητα. Και αυτό είναι το σχέδιο επί του οποίου θα στηριχθεί η κατασκευή. Δεν λέμε ότι είναι απίθανο, αλλά δεν είναι αδύνατο, αλλά είναι απίθανο να συμβεί κάποιο πρόβλημα. Ο σχεδιασμός λοιπόν θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την, το ενδεχόμενο της σεισμογενούς δραστηριότητας, αλλά η πιθανότητα να συμβεί κάτι σοβαρό με βάση τις αναλύσεις μας ε, ε, είναι εξόχως απίθανη. Ε, γι' αυτό αυτό που είπα δεν είναι σε αντίφαση. Ένα τελευταίο σχόλιο τώρα σε σχέση με τις δηλώσεις της κυρίας ακτιβίστριας. Δηλαδή πώς φτάνουμε στο 75% των ανθρώπων που αντιτάσσονται δεν το ε, ξέρω εγώ και γι' αυτό δεν μπορώ και να το σχολιάσω. Στη δική μου χώρα ποτέ η κυβέρνηση δεν οργάνωσε δημοψήφισμα για την πυρηνική ενέργεια. Γιατί ακριβώς οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η κοινή γνώμη θα οδηγούσε σε διαφορετικές επιλογές. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θεώρησα τη συζήτηση που προηγήθηκε ιδίως ενδιαφέρουσα. Ασχοληθήκαμε με πολλά θέματα, θέματα τα οποία θα οδηγήσουν ίσως και σε διαφορετικές πρωτοβουλίες, ιδιαίτερα με τη νέα κυβέρνηση που θα ακολουθήσει τις εκλογές της 12ης Ιουνίου. Η επόμενη συνεδρίασή μας θα γίνει λοιπόν στις 15 Ιουνίου. Θα προσπαθήσουμε να αποκρυπτογραφήσουμε τα αποτελέσματα των εκλογών που θα έχουν γίνει τρεις μέρες πριν. Ευχαριστώ όλους λοιπόν που πήραν μέρος στη συζήτηση. Ευχαριστώ για την παρουσία της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που παρουσίασε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η συνάδελφος από την Κωνσταντινούπολη δεν μας ακούει πια. Σας ευχαριστώ όλους. Θα συναντηθούμε στις 15 Ιουνίου. Γεια σας.